La seduta è aperta. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Άντερσον για διαδικαστικό. You have the floor. Έχετε το λόγο. Άντερσον, you have the floor. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι ήταν δύσκολη η απόφαση, αλλά ήθελα να πω σήμερα ότι η απόφαση για καθυστέρηση της ψηφοφορίας για τη δικιά μας τουλάχιστον αντιπροσωπεία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πώς το εκλαμβάνουν οι πολίτες της Ευρώπης. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη για αυτό το θέμα.